Κυρίε oh, euh, and gentlemen. και κύριοι, καλώ ήρθατε στη συνάντηση συνεδρίαση αυτή τη κοινοβουλευτική μα Επίτροπή, Θα ξεκινήσω με τι αναγγελίε Προέδρου. Thank Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λοιπόν, οι συντονιστές έλαβαν τις εξής αποφάσεις και αποφάσισαν ως εξής. Η κυρία Φεράρα διορίζεται η συγγήτρια για το αίτημα της άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κυρίου Σωτηρίου Ζαριανόπουλου η κυρία Ρέγνερ τώρα στη συνέχεια διορίζεται η συγγήτρια για το αίτημα άσυσης κοινοβουλευτική ασυλία του κυρίου Θεοδόρου Ζαγοράκη. Ο κύριος Χρυσόγονος στη συνέχεια διορίζεται εισηγητής για το αίτημα άσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κυρίου Γιάννου Σκόρβιν Μίκε. Ο κύριος Καβαντά στη συνέχεια διορίζεται εισηγητής για τη γνωμοδότηση για τις διαδικασίες και πρακτικές που αφορούν ακροάσεις επιτρόπων, υποψήφιων επιτρόπων και μαθήματα που πρέπει να συναχθούν από τις διεργασίες του 2014 όπως ακολουθήθηκαν. Η κυρία Κάουφμαν διορίζεται εισηγήτρια για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών οι συντονιστές συμφωνούν στη συνέχεια να προταθεί μια προφορική ερώτηση για την επικύρωση της σύμβασης του Μαρακές. Θα διανεμηθεί ώστε να εγκριθεί μέσω γραπτής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Προτάσεις ψηφίσματος από πλευράς Άλτο Πατριτσέλο και Μαραμπιζότο σημειώθηκαν και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 141 εγκρίθηκαν, υιοθετήθηκαν, θα διανεμηθούν και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της κοινοβουλευτική μας Επιτροπής. Μια κρόση για την ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών όσον αφορά τα, ε, νομικά, τα, δικαστικά επαγγέλματα θα προχωρήσουν ώστε να ζητηθεί και μία μελέτη που θα ζητήσουμε να εκπονηθεί. Μετά από την εκπόνηση αυτής της μελέτης θα δούμε ποια συνέχεια θα δοθεί. Η κυρία Χάουταλα θα προετοιμάσει ένα έγγραφο εργασίας και με μία πρόταση για κανονισμό και διοικητικές νομικές διαδικασίες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η κυρία Χάουταλα θα αναφέρεται σε ομάδα εργασίας που θα συντίθεται από, άτομα, από ένα άτομο από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Οι εξή νομοθετικές πρωτοβουλίες για εκθέσεις θα προχωρήσουν κοινέ προδιαγραφές για τις αστικές υποθέσεις, προστασία ευάλωτων ενηλίκων, διασυνοριακή αναγνώριση θεμάτων υιοθέτησης, περιορισμός περίοδου όσον αφορά οδικά τυχήματα και για τις διαδικασίες αυτές η κυρία Ντέλεβο θα είναι η εισηγήτρια. Δεν έχουμε ακόμα τους υποψήφιους εισηγητές για τα υπόλοιπα εκκρεμούντα θέματα. Η κυρία Ντέλεβο λοιπόν θα προταθεί ώστε να είναι μέλος στην ε, ΣΤΟΑ. προτάσεις ε, για τα προγράμματα και σχέδια ΣΤΟΑ ζητούνται. Το πρόγραμμα έρευνας ε, επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται και μία μελέτη για την ε, εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διάφορα επαγγέλματα και μία μελέτη για την εφαρμογή, δικαστική εφαρμογή θεμάτων οικογενειακού δικαίου. Και έτσι θα μπορέσουν να ενταχθούν υποψήφοι στην ομάδα επαϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων και θα δοθεί συνέχεια στη συνέχεια. Έτσι το Ίδρυμα ε, Κοινοτικού Δικαίου θα κάνει παρουσίαση στην, στην Επιτροπή μας στις 16 Απριλίου για το ELI εγχείρημα σε σχέση με τις ε, ε, διακρατικές αρχές ε, για τις αστικές υποθέσεις. Ο πρόεδρος θα συντάξει ένα μη έγγραφο, non-paper, για την διαπραγμάτευση μεταξύ, σε σχέση με μια νέα διοργανική συμφωνία για καλύτερη νομοθετική δραστηριοποίηση και έργο και θα υποβληθεί στους συντονιστές η πρόταση. Τελευταίο θέμα, η θα μεριμνήσει η Επιτροπή μας να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στις διάφορες αυτές υποθέσεις. Αυτά είναι τα θέματα επί των οποίων έλαβαν αποφάσεις οι ε, συντονιστές. Και ακολουθώντας τώρα το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής μας για το σημείο 11 το οποίο δεν καλύψαμε χτες και θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Κοφεράτη που δεν, βρίσκω δεν βλέπω να, να παρίσταται. Η κυρία Ρέγνερ έχει λοιπόν τον λόγο σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω ε, τις απολογίες του κυρίου Κοφεράτη το συγγνώμη για την απουσία του που έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν μπορεί να παραστεί και μου ζήτησε να παρουσιάσω εγώ τα συμπεράσματά του και δεν, είναι, δεν θα είναι σε θέση να παραστεί σήμερα και έτσι θα προσπαθήσω εγώ να σας πω ευθύ αμέσω ποια είναι τα κυριότερα σημεία στα οποία έχει καταλήξει. Όπως γνωρίζετε η έκθεση του κυρίου Κοφεράτη παρουσιάστηκε στις 19, ε, κατατέθηκε στις 19 Ιανουαρίου. Εν τω μεταξύ αρκετά μεγάλος αριθμός τροπολογιών κατατέθηκε. 404 συνολικά τροπολογίες κατατέθηκαν από τους σκιώδεις εισηγητές αλλά και από άλλους συναδέφους ευρωβουλευτές. Η ψήφιση <clears throat> προβλέπεται να γίνει το Μάρτιο και αυτό σημαίνει ότι πολλά πρέπει να γίνουν και σε σχέση με τον κύριο Κοφεράτη και τους άλλους σχεώδεις εισηγητές που εμπλέκονται για να καλυφθεί αυτή η πρόκληση, αυτό το μεγάλο έργο, ώστε να γίνει η προσπάθεια να ξεβρεθούν και συμβαστικές προτάσεις. Τώρα, κατά το μάλλον ήτον, το θέμα είναι ποια συνέχεια θα δώσουμε σε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να υπάρξει στενή συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚΟΝ και να δούμε και το θέμα του άρθρου 54. Τώρα, σε σχέση με τα ίδια τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν υποστήθενται υποσυζήτηση. Το πρώτο κεφάλαιο της οδηγίας, όπως γνωρίζετε, αφορά την δυνατότητα εταιριών να ταυτοποιούν να, ε, ποιοι είναι οι μεριδιούχοι, οι ομολογιούχοι τους, ε, να διευκολύνεται η διάχυση αυτών των πληροφοριών για να, να ασκούν τα δικαιώματά τους τα άτομα αυτά. Οι θέσει των διαφορετικών πολιτικών ομάδων δεν ε, απέχουν ε, πάρα πολύ η μία από την άλλη και έχει την πρόθεση να εξευρεθούν συμβιβαστικέ λύσεις ο κύριος Κοφεράτη. Είναι σημαντικό ε, ο τρόπος και η διατύπωση αυτών των πληροφοριών όπως θα διαβιβάζονται να είναι εύληπτος και να είναι σαφής να υπάρχει ένα ισοδίκαιο πλαίσιο δράσης και δραστηριότητας και να μην υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα και εργαλεία από πλευράς κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Το επόμενο μείζον θέμα είναι ο μηχανισμός για να υποστηρίζονται τα θέματα των, της μακρόχρονης ε, ε, ιδιότητας μεριδιούχου ή ομολογιούχου. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τα άτομα αυτά μακρόχρονα ώστε να υπάρχει αηφορία που θα διασφαλίζεται, ώστε ε, οι διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες να διασφαλίζονται. Έχει μεγάλη σημασία να υιοθετούν τα κράτη-μέλη τους αντίστοιχους αναγκαίους μηχανισμούς, ώστε να καλύπτονται τα ζητήματα αυτά και να διασφαλίζονται επαρκώς. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα λοιπόν, όπου ο κ. Κοφεράτη θα προσπαθήσει να εξεύρει συμβιβαστικές λύσεις που θα προτείνει. Ένα από τα φλέγοντα θέματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι ο ορισμός της, ε, της αναλογίας που πρέπει να διέπει τα μερίδια και τις ομολογίες. Εδώ υπάρχουν διάφορες, διαφορετικές αρχές. Κάποιες από τις μείζονες αρχές πρέπει να, να διασφαλίζονται. Ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές τάσεις σε σχέση με τις τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό για τον κύριο Κοφεράτη λοιπόν αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διασφαλιστεί και να συνεχίσει να υφίσταται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή που θεωρεί ότι θα είναι δεσμευτική η ψήφιση και η διασφάλιση όσον αφορά την πολιτική σε σχέση με τις αμοιβέ ε, και τις, ε, τα, τα ποσά τα οποία θα ε, καταβάλλονται. Είναι λοιπόν πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή και θα την αντιμετωπίσει ο κύριος Κοφεράτη. Το ένα θέμα είναι η διασφάλιση της διαφάνειας σίγουρα και το άλλο θέμα είναι ο μηχανισμός που θα προτείνεται να μην αντιβαίνει όποιες, οποιαδήποτε από τα συστήματα της αρχές ε, της εταιρικής διαχείρισης που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Και όσον αφορά τις ε, συναφείς δραστηριότητες, ε, οι τροπολογίες που έχουν τεθεί από διάφορους συναδέλφους θέλουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα θεσπιστεί που θα είναι πιο ευέλικτο από εκείνο που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να είναι φιλόδοξος ο τελικός στόχος και να διασφαλίζει ένα πλαίσιο αποτελεσματικότητας. Αρχές που πρέπει να διασφαλίζουν ένα εύθετο επίπεδο ελέγχου που θα επιτυγχάνεται επ' αυτών των συναλλαγών. Και όπως είπα και πιο πριν, με ένα υψηλότερο βαθμό διαφάνειας οπωσδήποτε όλα αυτά. Τελευταίο εξίσου σημαντικό, αρκετές διάφορες πολιτικές ομάδες ε, προτείνουν να υπάρξει υποχρέωση αναχώρα να υποβάλουν εκθέσεις όσον αφορά ε, μεγαλύτερες εταιρείες ε, που εμπλέκονται εδώ. Σε σχέση με την οδηγία για τη διαφάνεια κατά την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία όπως ε, το είχαμε προωθήσει αυτό ε, στο θεματολόγιο μας ε, είχαμε προαγάγει το θέμα και έτσι υποστηρίζει λοιπόν αυτές τις αρχές ο κύριος Κοφεράτη και προσβλέπει στην περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων αυτών με τα μέλη της Επιτροπής. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας που προσέξατε τα όσα σας ανέφερα από τον κύριο Κοφεράτη. Ευχαριστώ πολύ και τότε Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες. Αυτές καταδεικνύουν ότι προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για τη νέα αυτή οδηγία, η οποία τελικά θα επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας πάρα πολλών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι 487 τροπολογίες καταδεικνύουν ε, ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από μια συμφωνία, άρα πρέπει να καταβληθούν πάρα πολλές προσπάθειες τις επόμενες εβδομάδες για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εξυγχρονίσουμε μια οδηγία δημιουργώντας ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να εμπλέξουμε περισσότερο τους μετόχους τη διακυβέρνηση των εταιριών. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιβαρύνουμε οικονομικά και διοικητικά τι επιχειρήσει. Σιγά σιγά βγαίνει από την κρίση, την απέσια αυτή κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κρίση η οποία βάρινε πάρα πολύ τον επιχειρηματικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να ενισχύσουμε το βιομηχανικό τομέα προκειμένου πραγματικά να ανακάμψει η οικονομία. Πρέπει να προωθήσουμε την την εργασία των επιχειρηματιών, δεν θα πρέπει να τους βαρύνουμε με νέα κόστη, με νέα διοικητικά άκθη και θα πρέπει να καταφέρουμε να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική. Θα πρέπει οι ιδιωτικές εταιρείες να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα στα πλαίσια μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Κάθε, κράτο, κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανόνες, το δικό, το, το, τα δικά του, το δικό του μοντέλο. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε εμείς ένα μοντέλο μοναδικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, θα πρέπει ο κύριος Κοφεράτη, μόλον ότι εμείς έχουμε κάποιες αμφιβολίες και μια κάποια δυσπιστία για κάποιες προτάσεις, να καταλήξει μαζί μας σε μία καλή λύση για όλες τις επιχειρηματίες. Για Έχουμε πολλά προβληματικά σημεία. Πρώτον, θέλουμε όντως να μπορούν οι επιχειρήσεις να εξακριβώνουν ποιοι είναι οι μέτοχοί τους. Κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένας πιο ανοιχτός διάλογος με τους μετόχους και μια πιο βιώσιμη ενεργό συμμετοχή τους. Όμως δεν θα πρέπει αυτό να γίνεται από ενδιάμεσους, αν αυτό δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να έχουν οι ίδιες επιχειρήσεις χωρίς να απευθύνουν αναγκαστικά σε ενδιάμεσους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι αποδοχές των διευθυντών, των διοικητικών στελεχών η πρόταση που γίνεται εδώ πέρα, να περνάει δηλαδή η απόφαση αυτή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είναι πραγματικά συζητήσιμη. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να προκύψουν εδώ πέρα πολλά προβλήματα και να έχουμε μάλιστα και διακριτική μεταχείριση, να μην έχουμε δηλαδή μία αμερόληπτη αντιμετώπιση. Νομίζω ότι οι επιχειρήσει μόνε του θα πρέπει να καθορίσουν και όχι περνώντα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ποιε θα είναι οι αποδοχέ των διευθυντών. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να προσελκύσουν του πιο άξιου διευθυντέ. Επίσης η πρόταση που ζητά από τους εκπροσώπους των εργαζομένων να μπορούν και αυτοί να αποφαίνονται για την, ε, τις αποδοχές των εργαζομένων είναι μια πρόταση που δεν μας βρίσκει σύμφωνο. Θεωρούμε ότι θα είναι εντελώς αντιπαραγωγική. Επίσης, ε, οι σχέσεις με τα στεδεμένα μέλη. Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις πάλι θα πρέπει από μόνες τους και θελούσια να μπορούν να επιλέγουν με ποια στεδεμένα μέλη θα συνεργάζονται και δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να επιβάλλουμε εμεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, στα πλαίσια των Διοικητικού Συμβουλίου μπορούμε να έχουμε ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Μπορούν τα στεδεμένα αυτά μέλη όντως να βοηθήσουν στην καλύτερη αξιολόγηση της λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά δεν μπορούμε εμείς να έχουμε μία υποχρέωση προς αυτό. Τώρα, άνω του 5% ε, των ε, λειτουργικών των συναλλαγών μιας επιχείρησης είναι συναλλαγές με σταταμένα μέρη. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί. Αν διατηρηθεί με τον τρόπο που προβλέπεται αυτή τη στιγμή στο κείμενο, θα βγει σε πάρα πολλές καθυστερήσεις... καθώ επίση και σε ιδιαίτερα ψηλό για τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει απλώς να προβλέπουμε ε, συγκεκριμένου κανόνε για τι συναλλαγέ με τα στεδεμένα μέρη, θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα μητρό που να βλέπουμε ακριβώ ποια είναι τα στεδεμένα αυτά μέρη τα οποία συνεργάζονται με τι επιχειρήσει. Η συνέλευση αυτή επίση των ε, μετόχων, ο τρόπο με τον οποίο περιγράφεται στην έκθεση αυτή δεν συνάδει με το ζήτημα τη εμπιστευτικότητα που θα πρέπει να υπάρχει όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία συζητώνται πολλέ φορέ στα πλαίσια των ε, γενικών συνελεύσεων των μετόχων θα πρέπει η επιχείρηση, ένας επιχειρηματικός όμιλος να μπορεί να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητε που του δίνονται κάθε φορά που συνεργάζεται με στεδεμένα μέρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και βλέπετε ήδη από την παρέμβασή μου αυτή ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία επί των οποίων καλούμε θα εργαστούμε ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Καβαντά. Πρόεδρε. Στον κύριο Κοφεράτη να αποστείλουμε ευχαριστίες, διότι το έργο του είναι πολύ σχηδές και σε βάθος. Χαιρόμαστε που ασχολήθηκε με το θέμα ο κύριος Κοφεράτη. Συμφωνούμε με πολλά σημεία, με άλλα βεβαίως διαφωνούμε. Θα ήθελα να πω ότι το ρύθμα πλέον για μας είναι κατά πόσον πρέπει να θέσουμε όρια στον χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό που έκανε τη ζωή δύσκολη σε πολλές επιχειρήσεις, που αποσταθεροποίησε πολλές από αυτές ή αν πρέπει να ευνοήσουμε τον ε, οικογενειακό επιχειρηματικό καπιταλισμό όπως τον ζούμε στη Γερμανία που δείχνει την σταθερότητά του. Το έργο λοιπόν αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί βεβαίω. Πρώτον ω προ ε, τι ε, τροπολογίε και τι εκθέσει αναχώρα. Εδώ είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα. Με την εξή έννοια. Εάν πάρουμε τι τροπολογίες κατά γράμμα θα υπήρχαν αρνητικέ επιπτώσει για χώρε και για επιχειρήσει και από αυτήν την άποψη θα πλήταμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η μονομερής δημοσιοποίηση πληροφοριών στις ε, αναχώρα εκθέσεις αποτελεί στρατηγικό λάθος, λάθος στρατηγικής. Αποκαλύπτοντας τέτοιου είδους πληροφορίες, που είναι ευαίσθητες πληροφορίες, ρίχνουμε νερό στον μήλο των φορολογικών αρχών σε αναδείμενε αγορέ και έτσι θα μπορούσαμε να θέσουμε σε κίνδυνο ακριβώ αυτέ τι επιχειρήσει, οι οποίε θα καλούνται να πληρώσουν δύο φορέ φόρο. Αυτό εννοείται ότι θα είχε αρνητικέ επιπτώσει την κερδοφορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και έτσι θα στερούνται ορισμένα κρατημέλη μελη φορολογικών εσόδων στην επικρατή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μιλήσω καν για το πόσο θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Όλα αυτά θα δυσκόλευαν πάρα πολύ τις διαδικασίες και βέβαια θα είχαμε την δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών, εμπορικών μυστικών μεταξύ άλλων, κάτι το οποίο και πάλι θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίων αγοράς εκτός των συνόρων μας. Είναι βέβαια πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε όταν ε, έρθει η ώρα για το εμπορικό απόρριτο. λοιπόν μία μελέτη αξιολόγηση επιπτώσεων πριν περάσουμε στις αναχώρα εκθέσεις. Εάν θα χρειαστούν αναχώρα εκθέσεις μετά από την αρχική μελέτη, τότε θα προσπαθήσουμε εμεί να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις, ζητώντας την εφαρμογή όλων αυτών σε επίπεδο G20. Δύσκολο βεβαίω, δεν το βλέπω. Απόκλειδες πάντως καταρχήν σε κάθε περίπτωση την διπλή φορολόγηση. Έτσι ώστε τουλάχιστον να περιοριστούν οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες, τα απολύτως απαραίτητες, τις απολύτως απαραίτητες για τις ε, φορολογικές διοικήσεις των χωρών. Αυτά ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι η οδηγία για τα δικαιώματα αυτών των ομολογιούχων ξεπερνά τον ε, στόχο που έχουμε θέσει όταν ασχολείται μόνο με το θέμα του πώς μπορεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα επιχειρησιακές τέτοιες δραστηριότητες να καλύπτονται. Θα λέγα ότι αυτό αν γίνεται επαρκεί πλήρως, αλλά εδώ υπάρχουν πάρα πολλές πτυχέ που ξεπερνούν όμως αυτό το πλαίσιο και πρέπει να πω δεν είναι παντού αναγκαίο να γίνεται αυτό. Στο άρθρο 3α έχουμε αυτήν την ε, ταυτοποίηση των ε, ε, ομολογιούχων και θα πρέπει να είναι σαφές ε, πώς λειτουργούν τα πράγματα και μπορεί να, συναχθεί η σύνδεση με τα εθνικά υφιστάμενα συστήματα. Δεν πρέπει όλα να γίνονται με καινούριο νέο τρόπο και τα εθνικά συστήματα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη όσα έχουν με ονομαστικές μετοχές και σε σχέση με αυτές τις ε, ονομαστικές μετοχές ε, μέσω του μητρώου ε, μετόχων μπορούν, να ρυθμίζονται αυτά τα θέματα. Δεν πρέπει να θέσουμε πληθώρα νέων καθηκόντων. Και για το κόστος των διαμεσολαβητών, των μεσολαβούντων, πάλι από τις επιχειρήσεις καλύπτονται αυτά τα κόστη σε σχέση με το κύριο συμφέρον που έχουν να εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σε σχέση με τις εκτελεστικές ε, πράξεις ε, υπάρχει μεγάλο δυναμικό πολύ μεγάλη υπερβολική γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους επιβάρυνση όταν όλα με σαφήνεια καθορίζονται σε μια τέτοια οδηγία και όταν και τα εθνικά συστήματα λαμβάνονται υπόψη και συνδέονται με αυτήν. Και σε σχέση με την ρύθμιση για το 9α και το 9β για τις αμοιβέ και την έκθεση για τις αμοιβέ. Πιστεύω ότι ε, αποδυναμώνεται το εποπτικό ή διοικητικό συμβούλιο ή όταν μετατίθεται αυτή η αρμοδιότητα αλλού και υπάρχει διάρρηξη του διοικού συστήματος ε, ας το διατυπώσω έτσι. Τίθεται επιπρόσθετα το ερώτημα της ευθύνης Ποιος ευθύνεται, το Διοικητικό Εποπτικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις του όσον αφορά το πλαίσιο των αποφάσεών του για τις αμοιβέ. Θα ε, δημιουργείται όμως ε, μεγάλο κενό αν ρυθμίζαμε κάποια θέματα και σε σχέση με την ευθύνη απολύπαμε κάποια, ε, εξαιρούσαμε κάποια θέματα. Γι' αυτό η πολιτική αμοιβών σε αυτή την πρόταση στο σημείο 9α για το ευρωπαϊκό επίπεδο το θεωρώ κάτι ανέφικτο να λειτουργήσει σωστά. Και μετά το σύνολο της αμοιβή, ε, όπως αναφέρεται, ε, θα περιόριζε σημαντικά την επιχείρηση στην ευελιξία της όσον αφορά την ελαστικότητα που απαιτείται. Και για το 9Γ η έγκριση της ε, ε, συνέλευσης των μετόχων ε, νομίζω και πάλι εδώ προβλέπει η ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την ρύθμιση ε, αυτών όλων των θεμάτων, αυτή η ρύθμιση όλων αυτών των θεμάτων θα επιβάρυνε πολύ γραφειοκρατικά το πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Και τα θέματα συνέλευσης μετόχων θα μας οδηγούσαν στο να χρειαζόμαστε σαφέστατες, σαφέστατους ορισμούς ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο διαφάνειας όπως απαιτείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν ζήτησε τον λόγο. Συμφωνούν οι βουλευτέ. Να δώσουμε τον λόγο στην Κομισιόν. Ωραία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν ευχαριστεί θερμά τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έργο τους επί της πρότασης της Κομισιόν, της προτινόμενης οδηγίας. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες προς ε, διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι καλό που παραμένετε φιλόδοξοι, δεν θέλουμε να χάσουμε την προσθεμένη αξία της οδηγίας, αυτός είναι και ο στόχος μας και αυτό έχουμε στο μυαλό μας και θα έχουμε στο μυαλό μας να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Πιστεύουμε ότι απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας. Τα προτείνομενα στην οδηγία μέτρα είναι μάλλον ήπια είναι μάλλον ε, γενικόλογα. Οπότε όπου είναι να γίνουν αλλαγές, να γίνουν, αλλά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της οδηγίας. Χρειάζονται επίση διαδικαστικές εγγύησεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, αμοιβέ των διαφορών εμπλεκομένων και συνδεμένων μερών. Δεν πρέπει επίση να μειώσουμε περιβολικά την ενημέρωση των μετόχων. Δεν θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να προσελκύσουμε παιδιτές και δι μειοψηφία. Τα σχετικά μέτρα λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέροντα σε δύο επίπεδα απτώνται πολύ τεχνικών ζητημάτων που δεν μπορούν να συζητηθούν επαρκώς στο επίπεδο 1. Απερούνται όμως για την ορθή εφαρμογή των κανόνων στο επίπεδο 1. Οι επιχειρήσεις βλέπουμε ότι υποστηρίζουν την τυποποίηση και οι επιχειρήσεις και οι ενδιάμεσοι και οι επενδυτές. Και υπάρχουν και άλλα σημεία στην οδηγία. Όσον αφορά τα επιπλέον κίνητρα για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Θέλουμε φυσικά να τους ενθαρρύνουμε, όμως ορισμένοι από τους προτινόμενους μηχανισμούς οδηγούν προς τα αποτέλεσμα, διπλά δικαιώματα ψήφου για παράδειγμα. Εμείς θα θέλαμε να ευνοήσουμε τους ε, μετόχους πλειοψηφίας, αλλά δεν θέλουμε να αποκλείσουμε τους μετόχους μειοψηφίας. Θέλουμε να ωφελθούν και αυτοί. Συνεπώς χρειάζεται αξιολόγηση επιπτώσεων, πιο προσεκτική. Η Κομισιόν αυτά ακριβώς εξετάζει αυτή τη στιγμή. Φέτος θα γίνει μια δημόσια διαβούλευση και θα συντάξουμε έκθεση όσον αφορά την υπεύθυνη επένδυση. Και εξετάζουμε, όπω είπα, και τα κίνητρα για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Τώρα, όσον αφορά τις αναχωρά εκθέσεις, κατανοώ τις ενισχύσεις πολύ καλά όσον αφορά τη φορά αποφυγή, όμως ε, δεν είναι αυτό το κείμενο το κατάλληλο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Προσβλέπουμε φυσικά σε διαπραγματεύσει με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα. Να σα ενημερώσω επίση ότι η Κομισιόν για το θέμα τη φοροαποφυγή θα συνεχίσει το έργο τη βάσει των προτεραιοτήτων στο πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν για το 2015. Επίση, πρέπει να σταθμίσουμε πολύ προσεκτικά τι επιπτώσει τροπολογιών όσον αφορά τι αναχώρα εκθέσει, διότι ο διοικητικό φόρτο για τι επιχειρήσει μπορεί να είναι υπέρμετρα δυσανάλογα μεγάλος. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή όταν θα σταθμίσουμε τις τροπολογίες. Είμαι βεβαία ότι θα συζητήσουμε επικοδομητικά, με ειλικρίνεια, προς το κοινό καλό και εννοείται ότι παραμένω στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Ευχαριστώ. Κύριος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ισχυώδης συγητής για τους πρασίνους. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να πω κάποια πράγματα. Πρώτον, στα πλαίσια της ε, Επιτροπής μας. Θα μπορούσαμε να είμαστε και ευγενικοί. Μπορούμε να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Ζω Μαρή Καβαντά γιατί είναι σήμερα τα γενέθλιά του, έτσι δεν είναι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και το χρόνια πολλά, μόλον ότι ε, δεν συμφωνώ με ορισμένα από τα πράγματα τα οποία είπε. Λοιπόν, ήμουν ευγενικό στην αρχή, αλλά θα ήθελα τώρα να περάσω σε κάποια θέματα ουσία. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε ότι πρέπει να είναι κανεί πάρα πολύ επιφυλακτικό κάθε φορά που του γίνεται κομπλιμέντα. Γιατί ξεκινάει κανεί με κομπλιμέντα και στη συνέχεια προχωρά σε πιο αυστηρέ παρατηρήσει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό Ξέρω ότι υπόθηκαν ήδη πολλά πράγματα όσον αφορά τι αναχώρα εκθέσει καταρχά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη. Το είχα πει και την τελευταία φορά, το παραλαμβάνω και τώρα. Ο κύριο Κοφεράτη έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία. Έχει προσπαθήσει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμβαστική λύση. Πρέπει λοιπόν αυτό να το προγραμμίσουμε. Κύριε Καβαντά, εσεί μα είπατε ότι όσον αφορά τι αναχώρα εκθέσει, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να είχαμε αρχικά μια μελέτη αντικτύπου. Κοιτάξτε, τη μελέτη αντικτύπου την έχουμε στην πράξη αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο δισεκατομμύρια τα οποία αποτελούν αυτή τη στιγμή φοροδιαφυγή, τα οποία είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν τεχνικά ταμεία εξαιτία τη φοροδιαφυγή. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω μελέτη αντικτύπου. Δεν μπορούμε επίση να θελοτυφλούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε στα να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει επιγόντω να λάβουμε δράση και απέναντι στο πρόβλημα αυτό μπορούμε να απαντήσουμε με δύο τρόπου. Η πρόληψη και η καταστολή. Εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε προληπτικά μέτρα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε στα πλαίσια ενός κόσμου που επιβάλλει μόνο κυρώσεις και ποινές γιατί ουσιαστικά αυτό λειτουργεί ενάντια στι επιχειρήσει. Από την άλλη όμως, αν καταφέρουμε να έχουμε περισσότερα προληπτικά μέτρα, αυτό μας βοηθήσει να έχουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε δηλαδή την αδιαφάνεια που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Αναφερόμαστε για παράδειγμα σε ζητήματα όπως οι αποδοχές των διοικητικών στελεχών. Το ζήτημα αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό. Είναι εξίσου σημαντικό με το αν θα πρέπει τελικά να δηλώνουν τα πριμ τα οποία παίρνουν οι τρέιντερ, οι χρηματιστές του Λονδίνου ή όχι. Βλέπουμε όμως ότι ε, όσον αφορά την οικονομική κρίση υπάρχουν ζητήματα πολύ πιο σημαντικά από ό,τι αποδοχές των ε, διοικητικών στελεχών. Θα έλεγα ότι ένα από τα σημαντικότατα θέματα είναι η φοροδιαφυγή που αντιστοιχεί όπως σας είπα σε 2 δισεκατομμύρια. Επομένως ε, θα πρέπει και εσείς και εγώ όλοι μας να καταφέρουμε ο καθένας στη χώρα του να δημιουργήσουμε σύστημα ανάλογα με αυτό που ισχύει στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ απλό. Οφείλει κανείς να δηλώνει απλώς αυτά τα οποία χρειάζεται να καταβάλει στην εθνική φορολογία, στα εθνικά φορολογικά συστήματα. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό σε κάθε χώρα. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά για του επιχειρηματίε. Είναι πολύ σημαντικό για τι μεγάλε ιδίω επιχειρήσει να γνωρίζουμε ακριβώ ποια είναι τα χρήματα τα οποία καλούνται να καταβάλουν στα εθνικά φορολογικά συστήματα. Ξέρετε ότι πολύ συχνά οι μικρομεσαίε επιχειρήσει τι οποίε εκπροσωπούμε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιλέξουν φορολογικούς παραδείσους προκειμένου να φοροδιαφύγουν. Οι μικρές λοιπόν και μεσαίες επιχειρήσεις καταβάλουν σωστά τους φόρους τους η κάθε μία στη χώρα τους. Και δυστυχώς από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι καταφέρνουν να κερδοφορήσουν σε ορισμένες χώρες και στείλουν τέτοια φορολογικά συστήματα στη συνέχεια προκειμένου να μην καταβάλουν φόρους ή να καταβάλουν φόρους πολύ πιο χαμηλούς σε κάποια άλλη χώρα που έχει ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό σύστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσω των προτάσεων αυτών μπορούμε πραγματικά ουσιαστικά να βοηθήσουμε τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι εξίσου σημαντικό με το ζήτημα το οποίο θέσατε κι εσεί, Όσον αφορά δηλαδή τον βιομηχανικό τομέα, που όπως είπατε κι εσείς, ο βιομηχανικός τομέας όλο και περισσότερο πνίγεται από τις τάσεις που βλέπουμε στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κύριε Καβαντά λοιπόν, τη σήμερον ημέραν που ε, ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ μας λέει ότι δεν είναι πάρα πολύ περήφανος για το όσα έγιναν στα πλαίσια του Λουξ Leaks, αλλά έτσι συνέβαινε, μας είπε τότε, έτσι είχαν τα πράγματα. Ε, νομίζω ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή πρέπει πραγματικά να αλλάξει η κατάσταση, πρέπει πραγματικά να καταβάλλονται οι φόροι, πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά των επιχειρήσεων και θα πρέπει να έχουμε όλο και περισσότερη διαφάνεια και όχι αναγκαστικά μέτρα καταστολής. Αν ισχύσουν όλα αυτά, πραγματικά ο επιχειρηματικός κόσμος θα βελτιωθεί. Ο κύριος Καρίμ έχει το λόγο. Uh, thank uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μου πολιτική ομάδα είναι γενικά υπέρ των uh, στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν να κάνουν με τις βέλτιστες πρακτικές σε ορισμένα κράτη-μέλη, ιδίως αυτά που έχουν υψηλά πρότυπα όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Και θεωρώ ότι όντως θα πρέπει τα υψηλά αυτά πρότυπα να ισχύσουν σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εργαστούμε βάσει των προτάσεων της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως σε σχέση με την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ συχνά βέβαια αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ε, έχουμε μία πρόταση η οποία είναι κάπως ήπια, έχει να κάνει με το soft law, ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά η πρόταση αυτή να είναι πολύ πιο δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Πολλά προβλήματα βέβαια προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν υπάρχει αρκετή ευελιξία όσον αφορά τις βασικές αρχές που διέπουν την έκθεση. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες με κάποιες ιδέες παρεμβατικής φύσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αντικατοπτρίζονται άλλωστε και στις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει. Δεν συμφωνούμε με τα όσα λέγονται για τις απαιτήσει διαφάνειας. Οι απαιτήσει αυτές διαφάνειας έχουν να κάνουν με πολύ ευαίσθητες για τις επιχειρήσεις ε, πληροφορίες. Έχουν να κάνουν με ευαίσθητες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ουσιαστικά βάλουν κατά της ίδιας της τεχνογνωσίας και της εμπειρογνωμοσύνης των επιχειρήσεων. Καλούν οι επιχειρήσει να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις ε, οι οποίες ε, τελικά λειτουργούν αντίθετα με τους στόχους αυτής της οδηγίας. Επίσης δεν συμφωνούμε με τα όσα λέγονται για τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές τακτικές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και θεωρούμε ότι και πάλι αν δημιουργήσουμε μια εναρμόνιση των κανόνων για τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη τελικά θα επιβαρύνουμε περισσότερο τις επιχειρήσεις. Κατά την άποψή μας είναι σημαντικό να μην επιβαρύνουμε αρνητικά τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά την διοίκησή τους, όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες τις οποίες ε, παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές και δεν νομίζω πίσω ότι θα πρέπει να βάλουμε εμείς ενάντια στην θετική διαφορετικότητα που υπάρχει πολλές φορές στις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο εισηγητής κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες βαίνουν κατά των διαφορετικών παραδόσεων που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και γι' αυτό έχουμε εμεί υποβάλει τροπολογίες. Για παράδειγμα, η δημόσια γνωστοποίηση κάποιων πληροφοριών που δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να γνωστοποιούνται, κάποιες πληροφορίες που δεν αφορούν άμεσα τους μετόχους, τα γενικότερα συμφέροντα τα του ομολογιούχου ή τα όσα λέγονται για συγκεκριμένα κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δοθούν προς τους ομολογιούχους, αντί ουσιαστικά να προωθούνται άλλες προτάσεις που όντως θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ενεργό συμμετοχή των μετόχων. Η δική μου λοιπόν πολιτική ομάδα θεωρεί ότι όντως πρέπει να καταβάλουμε ακόμα πολύ περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να καταλήξουμε σε μια επικοδομητική συμβαστική λύση. Παρ' όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι Θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μία λύση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για τη δυνατότητα που μου δώσατε να εκφράσω την απόψή μου και να ευχηθώ και εγώ χαρούμενα γενέθλια στο ζώμα Καβαντά. Εδώ το γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά δεν έχει γεράσει καθόλου. Εγώ από την άλλη έχασα όλα τα μαλλιά μου όμως, όπως βλέπετε, και γενικά καταραίω. Πάντα. Κύριος Καβαντά έχει το λόγο. <laughs> Merci, Président. Merci. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Καρίμ. Αν έπρεπε να κεράσω σαμπάνια σε όσους μου εύχονται χρόνια πολλά σήμερα, θα κεραστευόμουν οικονομικά. Πρόεδρε, δύο λόγια για τον κύριο Τζιρά. Ξέρει πόσο τον εκτιμώ, αλλά εδώ τον εγκαλώ για παρανόηση των λόγων μου. Διότι γνωρίζετε ότι δεν είμαι και περίπτωση υποπτούς για υποστήριξη τη ε, φορολογική απάτη. Ήδη θα θυμάστε την έκκληση της Γενέβης το 1996 υπό τον εισαγγελέα Περτόσα ένας εξαιρετικό δικαστής θυμάστε η υπογραφή μου ήταν εκεί είχε υποστηρίξει την υπόθεση δεν ξέρω αν ήταν εκεί ήταν εσεί πολύ νέο αλλά έχετε υποστηρίξει την υπόθεση μαζί με την κυρία Βαζουλή Το λέω αυτό διότι είμαι αυστηρό, το ξέρετε. Και θέλω η Ευρώπη να έχει τη διάθεσή της τα μέσα για να δώσει την μάχη μαζί με Μεγάλη Βρετανία και Λουξεμβούργο κατά της φοροδιαφυγή που αποτελεί μάστιγα. Λοιπόν, θέλω να είμαι σαφής επί όλων αυτών. Δεύτερον, πρέπει οι αμοιβέ των μελών του ΔΣ να δημοσιοποιούνται. Γίνεται αυτό στην Αγγλία. Στην Ευρώπη ακόμα συζητάτε το θέμα. Έχουν γίνει βεβαίω κάποια βήματα προ την κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, εάν υπήρχε κάποια παρανόηση, σα να τα διευκρινίσω όλα αυτά για να τα ξεκαθαρίσω. Κύριε Ρέγνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πραγματικά για άλλη μια φορά, ιδιαίτερα, τον, τους από το ΕΛΚΑ, από την ΑΔΕ και ECR να μην κάνουν πάντα λόγο ότι ναι πρέπει κάτι να κάνουμε όπως λένε, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο φως στο σκοτάδι, περισσότερη διαφάνεια, αλλά από την άλλη πλευρά όταν πρόκειται για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων να λένε γιατί δεν θέλουν να ακολουθηθεί μια τέτοια πορεία δεν αισθάνομαι ιδιαίτερα ευχάριστα όταν βλέπω πολύ συγκεκριμένες χειροπιαστές προτάσεις που έχουν προταθεί που πάντα απορρίπτονται ως μη λέει ε, λειτουργικές από πλευρά τους. Ναι λένε για τη διαφάνεια αλλά όχι για τις χειροπιαστές δυνατότητες όταν πρόκειται για πληροφορίες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν κάτι να γίνει παραπέρα. Και όταν γίνεται μια συγκεκριμένη πρόταση δεν την δέχονται. Τώρα, σε σχέση με την αναχώρα έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν ένα θετικό μέτρο. Όλα αυτά τα πράγματα που σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές εκπονούνται, δηλαδή θέματα φοροαποφυγής, καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όλα αυτά να μπορέσουν να προχωρήσουν όμως με συγκεκριμένες προτάσεις. Η περισσότερη διαφάνεια φέρνει αρκετά στοιχεία και βλέπουμε ότι συγκλονίζονται οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης ότι πολύ γνωστές τράπεζες και μέλη διοικητικών συμβουλίων έχουν πάει τα χρήματά τους σε κάποιες χώρες όπου ισχύει το αφορολόγητο. Εδώ λοιπόν σε σχέση με τα θέματα αμοιβών πρέπει να επιτευχθεί πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια στην έκθεση Κοφεράτη αυτά αναφέρονται συγκεκριμένα. Δεν πρέπει λοιπόν να λέμε ότι ωραία έχουμε θετικούς στόχους που θέλουμε να επιτελέσουμε αλλά όταν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις να τις απορρίπτουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα παρακαλώ. Ναι ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι απαιτήσει για τη διαφάνεια και το πολύ σημαντικό στοιχείο της των εκθέσεων αναχώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατοχύρονται και τώρα έχει διασφαλιστεί σε σχέση με την συζήτηση και τους εμπλεκόμενους και με ιδιαίτερο τρόπο κιόλας. Ο κύριος από πλευράς Ντουράν αναφέρθηκε το θέμα της νομοθεσίας πρότυπο σε σχέση με τις προσπάθειές μας. Μια και βρισκόμαστε στην αρχή της νομοθετικής αυτής ε, ε, φάσεις για αυτό το ζήτημα πρέπει να οδηγηθούμε από αυτές τις προτάσεις και να ξεβρεθεί ο καλύτερος τρόπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουμε. Αν εγκαταλείψουμε αυτή την απέτηση τώρα, ε, τότε θα χωλαίνει το θέμα της εφαρμογής αυτού του πολύ σημαντικού στοιχείου, αυτής της πολύ σημαντικής αρχής. Εδώ θα ήθελα μια ιδέα να αναφέρω. Φυσικά οι εταιρείε πρέπει να ανταποκρίνονται σε πολύ μεγάλο αριθμό απαιτήσεων όσον αφορά εκθέσεις ε, που πρέπει να υποβάλλονται. Στο εγγύς μέλλον ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί ένα είδος κωδικοποίησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις απαιτήσει ε, για αυτές τις εκθέσεις, ώστε να έχουμε έναν εύληπτο, πιο απλό τρόπο, απλουστευμένο τρόπο σε σχέση με τα κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται σε σχέση με ε, ενιοποιημένες τέτοιες διατάξεις δεν γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή, ίσως όμως είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να επιτευχθεί σε μια επόμενη φάση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε έτσι τους, τον κατάλογο αγοριτών για αυτό το θέμα. Και μπορούμε να περάσουμε στο 15 τώρα, όπου θα έχουμε τις ψηφοφορίες. Πρώτα λοιπόν θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής ο ίδιος, ο κύριος Νεγκρέσκου, παρακαλώ. Ναι, Σε ευχαριστώ. Σε σχέση με την, ε, την παρέμβασή μου για το θέμα αυτό, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα ήθελα να πω ότι προσπαθήσαμε να γνωμοδοτήσουμε με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη η πρώτη γνωμοδότηση που είχε διατυπωθεί από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων κατά το παρελθόν. Να προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε κάποια στοιχεία τα οποία τονίζουν την ανάγκη να είναι πιο ανεξάρτητος ο φορέας αυτός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή και να είναι ανεξάρτητος όσον αφορά πολιτικές τάσεις και για το πώς ο διορισμός από πλευράς του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και των εντεταλμένων εισαγγελέων πώς θα γίνονται αυτοί οι διορισμοί καθώς επίσης και στοιχεία τα οποία αναφερόντουσαν τότε στην έκθεση που είχε συνταχθεί ε, στις νομοδοτήσεις ε, από πλευράς άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Επίσης προσπαθήσαμε από την άλλη πλευρά να αναφερθούμε και σε σχέση με το διασυνοριακό έγκλημα την ανάγκη δράσης και την ίση αντιμετώπιση όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά τα θέματα συζητήθηκαν από τους σκιώδεις εισηγητές. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συντάξουμε μια γνωμοδότηση που θα λαμβάνει υπόψη τις περισσότερες αυτές απόψεις και τα σημεία που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα και να ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε διανατάσεως των χειρών. Προχωράμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μετρήσατε. Πολύ καλά. Απορρίφθηκε τροπολογία, συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 8 υπέρ κατά να μετρήσουμε τι λέτε αποχές Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Έχετε τις κάρτες σας. Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε την 8. Τροπολογία 8 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, Δύο συνάδελφοι δεν έχουν βάλει τις κάρτες τους, δεν συμμετείχαν. Τώρα εντάξει. Ωραία. Η τροπολογία 8 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτής. I close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. Συγγνώμη, αποχές πρώτα. Μάλιστα, απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε, μάλιστα. Απορρίφθηκε. 11. Τροπολογία 11 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 13. Σε τμήματα. Όπως ζητήθηκε από τους σοσιαλδημοκράτες. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τι λέτε θα ελέγξουμε λοιπόν πρώτο τμήμα της 13 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα της 13 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 16. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τι λέτε. Ας ελέγξουμε όμω ηλεκτρονικά. Θα ελέγξουμε, ψηφίζουμε την 16, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε το ολογέ 18 σε τμήματα πάλι εδώ πρώτο τμήμα της 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα της 18 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 19 τώρα. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ωραία. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 σε τμήματα πρώτο τμήμα της 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα της 27 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος της 27 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας α, ένας δεν έχει συμμετάσχει ακόμα ωραία, πέρας ψηφοφορίας τώρα εγκρίθηκε τρίτο τμήμα της 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 28 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τι λέτε μάλιστα εγκρίθηκε εντάξει να σε ελέγξουμε ψηφίζουμε την 28 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας τώρα εγκρίθηκε λοιπόν πράγματι και τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης ως σύνολο. Το ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτού. Πέρας ψηφοφορίας. Λείπει ένας που δεν συμμετείχε. Μάλιστα, εγκρίθηκε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης ως σύνολο. Ε, we pass to... Και περνάμε στο σημείο 16. Εγκρισή σχεδίου έκθεσης με τη μορφή επιστολής. τέσσερι χειρός υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε κυκλισμένων των θύρων όποιος δεν δικαιούται συνεχίσει, παρακαλούμε να εξέλθει έτσι αυτές.